υπάρχουν και αντλίες θερμότητας που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε γιατί πρόκειται για την πεμπτουσία του μέλλοντος της ε, νέας εκβιομηχάνησης. Σας ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η κοινή συζήτηση. Η ψηφοφορία για τις εκθέσεις αυτές θα λάβει χώρα αύριο.